Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας συνεδρίαση. Πριν αρχίσουμε, θα πρέπει να σας ρωτήσω αν διαφωνείτε με τη ημερήσια διάταξη, αν έχετε καμιά αντίρρηση, όχι. Εγκρίνεται λοιπόν η ημερήσια διάταξη. We have a linguistic problem, unfortunate interpretation. Δυστυχώς ε, ε, δεν έχουμε διερμηνία σήμερα ούτε αύριο στα κροατικά και στα Ιρλανδικά. Κροατικά και γοδελικά. Ε, στη συνέχεια, ορισμός εισηγητών. Η Μάιτε Παγάσα Ορτουντούα ορίστηκε εισηγήτρια για επτά θέματα που εξετάζουμε μαζί για τις νέες ψυχοδραστικές ουσίες. Είναι πακέτο πάντως ε, και νομίζω καλό θα ήταν να διαπιστώσουμε ότι ε, έχει οριστεί η συγκήτρια για τα θέματα αυτά που εξετάζω όλα μαζί. Συμφωνείτε, ε, συμφωνείτε, συγγνώμη. Επίσης θα πρέπει να ανακοινώσω ότι αύριο ψηφίζουμε στις 10 η ώρα, ακριβώς 10 η ώρα, έχουν προβλεφθεί για αύριο οι ψηφοφορίε και βεβαιωθείτε παρακαλώ ότι θα έχετε μαζί σας τις κάρτες σας να ψηφίσετε. Επίσης, έχουμε και τα πρακτικά του Νοεμβρίου ε, και του Δεκεμβρίου του 2017. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις για τα πρακτικά αυτά, δεν διαφωνεί κανείς. Ωραία, εγκρίνονται τα πρακτικά. 13 Νοεμβρίου, 19 Οκτωβρίου, 10-12 Ιουλίου, 29-30 Μαΐου και του 17 όλα αυτά και 8 Ιανουαρίου του 2018. Σας καλωσορίζω λοιπόν στη δημόσια αυτή ακρόαση για την ε, ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Ξέρετε ότι η ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστίθεται με την υπηκότητα, την ηθαγένεια του κάθε πολίτη, δεν την υποκαθιστά και δεν την αντικαθιστά. Οι πολίτες της Ένωσης έχουν το δικαίωμα να κυλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα σε άλλα κράτη-μέλη, το δικαίωμα του εκλέγην και εκλέγεστε στις δημοτικές και τις ευρωπαϊκές εκλογές, την αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το δικαίωμα να προσφεύγουν στον Ευρωπαίο Μεσολαβητή, καθώς επίσης και το δικαίωμα να απολάβουν σε τρίτη χώρα της προστασίας των διπλωματικών και προξενικών αρχών κάθε άλλου κράτους μέλους. Η συνθήκη τη Λισαβόνα, η οποία υπογράφηκε το 2007, χορήγησε στου πολίτε τη Ένωση άλλο ένα δικαίωμα. Το δικαίωμα να ε, προχωρούν σε πρωτοβουλία πολιτών το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δήλωσε στο ψήφισμά του πρόσφατα στις 12 Δεκεμβρίου του 2017 ότι οι προσπάθειες για την προώθηση της ηθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνδέονται με την απόλαυση στην πράξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και με την ευκαιρία που δίδεται σε κάθε πολίτη να συμμετέχει στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης. Η έννοια της ηθαγένειας της Ένωσης ε, ήταν αφιλεγόμενη από τη δημιουργία της ήδη από τη συνθήκη του Μαστρίχτ σκοπός αυτής της δημόσιας ακρόασης είναι να ακουστούν εμπειρογνώμονες στο θέμα αυτό και τη σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων προκειμένου να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος της ηθαγένειας της Ένωσης στη ζωή των πολιτών αλλά και όσον αφορά το χώρο ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές ε, που ε, μας αφιερώνουν το χρόνο τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουν λάβει ήδη τις θέσεις τους ε, εδώ στο Προεδρείο. Θα ήθελα καταρχάς να δώσω το λόγο στον καθηγητή Δημήτρη Κοτσένοφ, ο οποίος είναι πρόεδρος του Τμήματος Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική ε, Σχολή στο Πανεπιστήμιο του Χρόνιγκεν. Θα είμαι πάρα πολύ αυστηρός με το χρόνο. 12 με 15 λεπτά έκαστος.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 Ε, η παρακαθήμενή μου, η κυρία Κωνσταντακόπουλος, έχει πολύ συγκεκριμένες απόψεις γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Οι βασικές ιδέες λοιπόν τις οποίες έχουμε μπροστά μας είναι ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν θα πρέπει να χάσουν το καθεστώ τους ε, ε, με τέτοιο τρόπο και ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα επιπλέον καθεστώς για τους Ευρωπαίους πολίτες οι οποίοι ε, τυχαίνει να ανήκουν σε μία, να είναι συνδεδεμένοι κατά κάποιο τρόπο με μια χώρα η οποία αποχωρεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε διάφορα επίπεδα ε, τίθεται το θέμα. Το πρώτο επίπεδο είναι πάρα πολύ απλό. Η δημοκρατία εδώ είναι κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία θα πρέπει να προσπαθήσουμε να σεβαστούμε την λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών σε επίπεδο κράτους μέλους και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι υποχρεωμένη να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε το άρθρο 4.2 στη συνθήκη, το οποίο <clears throat> υπογραμμίζει την σημασία των συνταγματικών παραδόσεων των κρατών μελών και αναφέρεται ακριβώς και στις ε, θεσμικές δομές των χωρών αυτών έτσι ώστε να διασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή του νόμου και σε εθνικό και σε υπερεθνικό επίπεδο. Κάθε δημοκρατία παράγει φυσικά νικητές και όπου υπάρχουν νικητές υπάρχουν και οι τιμένοι. Είναι σαφές λοιπόν ότι θα υπάρξουν και πλευρές που δεν θα είναι ικανοποιημένες από τη λειτουργία των δημοκρατιών στον κόσμο. Και αυτό <clears throat> μας απασχολεί σήμερα. Όλοι λοιπόν οι πολίτες της Ένωσης που χάνουν το καθεστώς τους, λόγω της λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών στην Ευρώπη είναι αυτοί οι οποίοι χάνουν σε επίπεδο δημοκρατικών δικαιωμάτων. Το θέμα το οποίο τίθεται λοιπόν είναι αν θα πρέπει να κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση και να δώσει κάποια επιπλέον δικαιώματα σε σχέση με τους πολίτες των τέος κρατών μελών. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα εδώ αν προσπαθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει ένα τέτοιο ρόλο Ιδιαίτερα σε νομικό επίπεδο αυτό είναι κάτι το οποίο θα οδηγήσει στην παραβίαση ακριβώς του συγκεκριμένου άρθρου του 4.2. Δεύτερον, το δεύτερο επίπεδο των προβλημάτων τα οποία δημιουργούνται από τις ιδέες του Φερχόφστατ είναι αν το καθεστώς αυτό επεκταθεί σε αυτούς που χάνουν την ευρωπαϊκή υπηκότητα, αυτό στην ουσία ε, αποστερεί από το άρθρο 50 οποιοδήποτε νόημα. Εν πάση περιπτώσει κάθε ρύθμιση που προβλέπεται από τις συνθήκες έχει, κάποια νόημα, έχει κάποιο νόημα, μπορεί να λειτουργήσει σωστά εφόσον το σύνολο λειτουργήσει σωστά. Και θα πρέπει να είναι φυσικά εφικτό το να εγκαταλείπει κάποιος την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δικαίωμα αποχώρησης είναι θεμελιώδες δικαίωμα της ιδιότητας του μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν αποσυρθεί λοιπόν η υπηκότητα από την εμβέλεια ακριβώς των εφικτών δυνατοτήτων μέσω των ειδικών αυτών μέτρων, αυτό είναι κάτι το οποίο φύγει ακριβώς το περιεχόμενο του άρθρου 50 και παράλληλα οι δημοκρατίες των μεμονωμένων χωρών ε, χάνουν τον ρόλο τους, το να καθοδηγούν δηλαδή και να οδηγούν σε αποφάσεις τους λαούς της κάθε χώρας χωριστά. Και ένα τελευταίο σημείο είναι ότι είναι προφανές το, το να ανοίξει ακριβώς μια συζήτηση για ένα νέο καθεστώς μετά το Brexit είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει προβλήματα σε επίπεδο ε, διαπραγματεύσεων, θα δημιουργήσει εμπόδια και θα δημιουργήσει και παράνομες καταστάσεις. Ένα επιπλέον σημείο, το τέταρτο σημείο σχετικά με τον Brexit. Να πω ότι η, αδίποτε, η ειδική μεταχείριση των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ηνωμένου Βασιλείου μετά τον Brexit θα στείλει ένα λανθασμένο μήνυμα σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει άμεσα μια μορφή αναλογικότητας και αμοιβαιότητας που απαιτεί το άρθρο 50. Μπορούμε να καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουν πολύ περισσότερα δικαιώματα από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο για αυτούς οι οποίοι πιστεύουν στην ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς λοιπόν, όσο και ελκυστική να είναι η ιδέα της διατήρησης των δικαιωμάτων αυτών των οποίων η χώρα αποχωρεί γιατί δημοκρατικά αποφασίστηκε η αποχώρηση αυτή ε, ταυτόχρονα είναι πάρα πολύ προβληματικό το να προσπαθήσουμε εμείς να αντικαταστήσουμε την εσωτερική δημοκρατία σε, χώρα, σε μια χώρα μέλος και να ακυρώσουμε το άρθρο 50. Και έρχομαι εδώ τώρα στην ιδέα της προστασίας των μειονοτήτων. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπερηφανεύεται ότι πραγματικά προστατεύει πάρα πολλά ευάλωτα ε, κοινωνικά γκρουπ, κοινωνικές ομάδες σε πάρα πολλά επίπεδα. Έχουμε ειδικέ οδηγίες για όλες τις μειονότητες. Προστατεύουμε τις εθνοτικές επίσης μειονότητες. Υπάρχει σημαντική νομολογία σε σχέση με την προστασία των μειονοτήτων θα μπορούσε να πει κανείς ότι η κατάσταση είναι σχεδόν ιδανική. Όμως υπό το φως της τελευταίας νομολογίας του Ευρωπαϊκού, της πρόσφατης νομολογίας, βλέπουμε εξελίξεις αρνητικές. Και θα τολμήσω να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πάρα πολλές φορές λειτουργεί σαν ένας φορέας, σαν ένα όχημα ε, προώθησης τυφλού εθνικισμού των κρατών μελών. Και αυτό γίνεται ακριβώς από την αναφορά την οποία έκανα το 4-2 της συνθήκης. Έχουμε κάποια τέτοια παραδείγματα δυστυχώς στις χώρες της Βαλτικής. Ας σας υπενθυμίσω λοιπόν πώς η προστασία των μειονοτήτων λειτουργεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πιο θα έλεγα δημοφιλές επίπεδο είναι απλά η εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης με βάση την προέλευση και την καταγωγή. Δεν τίθεται θέμα πλειοψηφία εδώ. Κάθε πολίτης που πάει σε μια άλλη χώρα, ναι μεν είναι τμήμα της ε, μειοψηφία, αλλά προστατεύεται απόλυτα. Και το ίδιο ισχύει επίσης ε, και με αυτούς οι οποίοι επιστρέφουν στις χώρες μέλη του. Με ε, χώρες μέλη Στην ουσία δηλαδή ε, απελευθερώνονται από τις απαιτήσει που υπάρχουν ε, για να μείνει κάποιος σε μια χώρα. Δεν χρειάζεται να γνωρίζει κανείς την τοπική γλώσσα, τις τοπικές μαγειρικές παραδόσεις, το να συμμετέχει στην λειτουργία των οργανώσεων, των κοινωνικών, πολιτικών κτλ. Είναι κάποιος καλοδεχούμενος ως έχει και είναι κάτι το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στο όνομα της συνταγματικής παράδοσης των κρατών μελών έχει αρχίσει να αφίσταται και ιδιαίτερα στην περίπτωση νομολογιών αποφάσεων των δικαστηρίων σε σχέση με την αντιμετώπιση των μειονοτήτων. Και αναφέρομαι στην περίπτωση Βεντρίν όπου η Λιθουανία της επιτρέπεται να συνεχίσει τις διακρίσεις εις βάρος της πολωνικής της μειονότητας ακόμα και σε μια περίπτωση όπου εφαρμόζεται πλήρως η ρύθμιση συνολική για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Έχει την δυνατότητα λοιπόν να κάνει εξαιρέσει ακόμα και στα πλαίσια της θεμελιώδους λογικής της ε, εσωτερικής αγοράς. Είναι πολύ απλή η λογική αυτή. Λέει ότι εφόσον ε, ε, εμπλέκεται αν θέλετε ε, σε επίπεδο διοίκησης τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς δεν υπάρχει διάκριση με βάση την εθνικότητα, την εθνότητα. Με βάση όμως την τελευταία απόφαση του δικαστηρίου, αν ανήκει κάποιος σε μια εθνότητα, το δικαστήριο λέω ότι κάποιες αντιμειονοτικές, εθνικιστικές, δικητικές παραδόσεις επικρατούν. Αποτέλεσμα είναι ότι στις βαλτικές χώρες οι μειονότητες Πολωνών, Εβραίων, Ρώσων, γιατί εδώ δεν γίνονται σεβαστές οι ρυθμίσεις της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών, δημιουργούν οι αποφάσεις αυτές ε, σε στερήσεις δικαιωμάτων. Δεν έχουν δικαίωμα να ονοματίζονται σαν παράδειγμα και υπάρχουν και άλλα επιπλέον μέτρα τα οποία δημιουργούν προβλήματα στην συγκεκριμένη περίπτωση. Η κατάσταση λοιπόν σε επίπεδο προστασίας των μειονοτήτων είναι τέτοια όπου η εσωτερική αγορά προστατεύει τους εκπροσώπους των πλειοψηφιών που πηγαίνουν σε διάφορες άλλες χώρες αλλά όταν πρόκειται όμως για τις εθνοτικές μειονότητες και τα μέλη τους δυστυχώς πάρα πολύ συχνά στερούνται ε, το καθεστώς της προστασίας των δικαιωμάτων λόγω ακριβώς του ιδιαίτερου ε, κατε, κατεξαίρεση ε, παραδοσιακού τύπου ρύθμισης που οδηγεί στον αποκλεισμό των μειονοτήτων ε, που κανονικά θα έπρεπε να τύχουν προστασίας. Και εδώ το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει, ε, θα έλεγα, λάβει εντελώς λανθασμένες αποφάσεις. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω εδώ αυτά τα οποία ε, έχει γράψει ο καθηγητής Μπόλκεν, ο οποίος λέει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί απέσιοι θεσμοί στον κόσμο, είναι το προθάλαμος της κόλασης, και αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να δούμε πότε οι θεσμοί αυτοί βλάπτουν την κατάσταση και στη συγκεκριμένη περίπτωση ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και στη συγκεκριμένη απόφαση ε, φοβάμαι ότι εγκαταλείφθηκε η προστασία της μειονότητας σε περίπτωση των βαλτικών χωρών και το δικαίωμα στο όνομα το εθνοτικό τώρα είναι κάτι το οποίο δεν έχουν οι μειονοτικοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά. Τώρα θα δώσω το λόγο στην ε, ε, κυρία Ντόρα Κωνστακοπούλου, καθηγήτρια Ευρωπαϊκού Δικαίου και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και Δημόσιας Πολιτικής από το Πανεπιστήμιο του Warwick. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε αξιότιμο μέλη της Επιτροπής συμμετέχοντες. Χαίρομαι που είμαι εδώ ε, για να μιλήσω για τη σχέση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ε, θα ήθελα να εστιαστώ ακριβώς σε αυτήν την ε, διασύνδεση και να αναφερθώ και στα θέματα, στα προβλήματα των μειονοτήτων. Με χαρά είδα ότι το προηγούμενο Δεκέμβριο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα σχετικό και ένα άλλο ε, ψήφισμα ε, πριν από μερικά χρόνια το οποίο αφορούσε ακριβώς ε, τις μειονότητες και ακριβώς σε αυτό το ψήφισμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητούσε ισχυρότερη διασύνδεση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εγώ πλήρως προσυπογράφω αυτήν την θέση και θα εξηγήσω για ποιο λόγο. Θα ξεκινήσω αναφερόμενη σε έναν ποιητή, τον Μάθιο Άρνο, το οποίος ε, έγραψε τα ποίηματά του 19ο αιώνα και ε, αυτός ο Μάθιο Άρνοτ μαθιο λοιπόν, αρνο όρισε πολιτισμό, τον πολιτισμό ως ε, τον εξανθρωπισμό του ανθρώπου στην κοινωνία και πίστευε ότι τα κράτη οφείλουν να εκπολιτήσουν και να εξανθρωπίσουν τα μέλη τους επιπροσθέτως όλων των άλλων. Καλή ψέων, των αναγκών των ανθρώπων ε, και επομένως ε, τι οι αυτές οι ανθρωπιστικές πολιτικές ε, και το αφήγημα περί ανθρωπισμού αποτελούν ακριβώς τα κεντρικά στοιχεία των πολιτισμένων κοινωνιών. Ωστόσο, στις συνθήκες Ευρατόμ και ΕΟΚ το 1957 δεν γίνεται κάποια αναφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά στη διάσκεψη κορυφή της Κοπενχάγης το τα νέα κράτη-μέλη εκείνης της εποχής ε, εξέφρασαν την πεποίθησή τους ότι οφείλουν να οικοδομήσουν μια κοινότητα δικαίου και δημοκρατίας ε, που θα ε, μετράει την και θα αντιμετωπίσει τις ανάγκες των μεμονωμένων ατόμων αλλά και της κοινωνίας μέσα στα πλαίσια των διαφόρων των διαφορετικών πολιτισμών. Ε, αργότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Στις ε, δεκαετίες που ακολούθησαν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καθώς και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά και με πολύ συνεκτικό τρόπο έτσι ώστε να δώσουν στα ανθρώπινα δικαιώματα κεντρική θέση εντός του νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, αρχικά, μέσω της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, έγιναν ε, τμήμα άρρηκτο των γενικών αρχών του Ευρωπαϊκού Δικαίου, καθώς επίσης και των πρωτογενών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέβαλε στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της ένταξης τους στο προσχέδιο ε, της ε, συνδικη Ευρωπαϊκής Ένωσης 17 Φεβρουαρίου 1984, καθώς επίση και με τη δήλωση περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών της 12 Απριλίου 1989 τροποποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2007, του 2007 ε, ε, αυτή η συνθήκη και έγινε νομικώς δεσμευτική ε, αφότου τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνα σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 της συνθήκης λειτουργίας και της δήλωσης υπαριθμών 1 του, του χάρτη ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, αναφέρεται δε σε απόφαση του δικαστηρίου ότι αυτή η, ε, αυτή χάρτα ε, αποτελεί την βάση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει νομική αξία για, την, για τις συνθήκες. Αναφέρεται δε ότι θέλουμε να ακολουθούμε την Ευρώπη η οποία βασίζεται στο δίκαιο. Επομένως και η, Ευρωπαϊκή, η, ηθαγένεια, η Ευρωπαϊκή οικογένεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν building blocks της ευρωπαϊκής ε, ταυτότητας και της έννοιας ε, του ευρωπαϊκού ανήκειν, του ανήκειν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, γνωρίζουμε βεβαίως ότι ε, ε, ε, στις αρχές του 1990 γίνεται η πρώτη ρητή αναφορά στις συνθήκες σε τέτοια θέματα. Αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι και αυτά τα δύο στοιχεία, δηλαδή από τη μία η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και από την άλλη, η από την άλλη τα θέματα των μειονοτήτων είναι εξαιρετικά σημαντικά. Ο A.G. Κόλομερ ανέφερε ότι Πώς είναι δυνατόν να αντιληφθεί κανείς ε, την ε, σχέση τους. Είναι γεγονός ότι και, τα δύο, ε, και οι δύο αυτοί θεσμοί έχουν ρητά αναγνωριστεί ήδη από την αρχή του, της δεκαετίας του 90. Ωστόσο θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν πιο σαφείς οι αναφορές. Πιο συγκεκριμένα ε, είναι γεγονός ότι η ευρωπαϊκή ε, ηθαγένεια μπορεί και πρέπει να ενσωματωθεί ε, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στα θεμελιώδη δικαιώματα. Ε, αυτή η σαφής διασύνδεση θα τους, ε, θα τους δώσει ε, μεγαλύτερη συνταγματική βάση και με τον τρόπο αυτό η έννοια του homo economicus θα μεταμορφωθεί σε homo civilaris. η κοσμοπολίτικη έννοια της ευρωπαϊκής ε, ε, ηθαγένειας ε, μπορεί λοιπόν να βρει την πλήρη της εφαρμογή σε αυτήν την διασύνδεση. Ο A.G. Κόλομερ θεωρεί ότι τα ε, δικαιώματα ε, που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια ε, συνδέονται βεβαίως με την έννοια της Ευρωπαϊκής Έννοιας αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει να αναφερθούν και στην αμοιβαία αλληλεξάρτηση. αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να μην σταθούμε μόνο σε αυτό. Θα πρέπει να υπάρχει και η νομική ε, διασύνδεση. Ε, βεβαίως ε, υπάρχουν πολλές, πολύ συχνά παραβιάσεις αυτών των αρχών όταν ας πούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνείται την αρχή της οικογενειακής επανένωσης ή δεν δίνει την πλήρη διακριτική ευχέρεια στα κράτη-μέλη να ε, έχουν κάποιες εξαιρέσεις όσον αφορά ε, την περιοχή της ηθαγένειας. Ε, βεβαίως θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και σε περίπτωση συλλογικών απελάσεων. Οι διασυνδέσεις και η εμβάθυνση της διασύνδεσης ανάμεσα στους δύο θεσμούς θα δώσει περισσότερες ευκαιρίες και στους δύο θεσμούς να ολοκληρωθούν. Ε, το άρθρο 7 ε, της ε, χάρτας ας πούμε αναφέρεται στην, στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής καθώς επίσης και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων στο άρθρο 8 και με τον τρόπο αυτό θα πρέπει, και θα πρέπει να βρεθεί ο τρόπος να διασυνδεθούν αυτές οι αρχές με τις διατάξεις που διέπουν την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Η απαγόρευση απαγόρευση των συλλογικών ε, ε, απελάσεων είναι ένα θέμα το οποίο επανειλημμένα έχει έρθει στο φως στη Γαλλία και στην Ιταλία λόγω των ε, υποχρεωτικών απομακρύνσεων των Ρωμά. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι περισσότεροι Ρωμά και στην Ελλάδα και στην Τσεχία και σε άλλες χώρες υφίστανται διακριτική μεταχείριση λόγω, της, λόγω του γεγονότος ότι ανήκουν σε αυτήν την εθνοτική ε, μειονότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει ότι ε, οπωσδήποτε για να συμπεριληφθούν τα δικαιώματα των Ρωμά στις, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριληφθούν δικαιώματα όπως είναι η στέγη, το δικαίωμα στην εκπαίδευση κλπ. Ε, βεβαίως ε, ε, η, η φυστάμενη διάκριση όσον αφορά ε, την στέγη, η ηγετοποίηση των Ρωμά εντός των Δήμων και των κοινοτήτων απαιτούν οπωσδήποτε δράση. Αλλά οι μελλοντικέ εξελίξεις της Ευρωπαϊκής Εθαγένεια θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ορισμένες από αυτές τις ανισότητες. Όλοι μπορεί να συμφωνήσουν ότι η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια έχει ε, την ε, δυνατότητα να δημιουργήσει, ε, να, να έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με πιο συγκεκριμένο τρόπο οι δομικές ανισότητες. Ας φανταστούμε ας πούμε ε, μια ευρωπαϊκή κοινοτική ηθαγένεια με σαφείς και ρητές αναφορές στην κοινωνική προστασία. Το ελάχιστο εισόδημα ε, για μια αξιοπρεπή ζωή. Την ε, προστασία την πρόσβαση στην ε, σέγη, στη στέγη, στην αντιμετώπιση ε, της ε, έλλειψης στέγης και την αντιμετώπιση των αστέγων, προστασία στην ασφάλεια στην εργασία, ας πούμε, δηλαδή μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θα ενσωματώσει τις αρχές του κοινωνικού πυλώνα. Ήδη από την, την δεκαετία του 1990 έλεγα ότι θα πρέπει οπωσδήποτε στο δεύτερο τμήμα της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής να υπάρχει μία αναφορά ε, στο ότι όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν την υποχρέωση να δείξουν αλληλεγγύη ε, σε ε, άλλους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε πολίτες τρίτων χωρών. Αυτή η υποχρέωση σημαίνει και προϋποθέτει σεβασμό στην αξιοπρέπεια των άλλων και απόρριψη οποιαδήποτε σε κοινωνικού αποκλεισμού και περιθωριοποίησης. Ε, και πιο ε, πρόσφατα ε, είπα ότι οι πιθανές υποχρεώσεις της κοινωνικής ηθαγένειας θα πρέπει να βρουν το δρόμο τους στις προβλέψεις και τις πρόνοιες μάλλον της ειδικής λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας που θα πρέπει στο μέλλον να σημαίνει καθήκον υποχρέωση όλων των κρατών μελών αλλά και της Ένωσης να προωθήσουν ισότητα των πολιτών πολιτών ε, επίσης ε, ε, την δυνατότητα να αντιμετωπιστεί η ένδια, η έλλειψη στέγης ε, και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Υποχρέωση επίσης από πλευρά των κρατών αλλά και της Ένωσης να προωθήσουν την ολοκληρωμένη και την συμπερίληψη όσον αφορά την πρόσβαση στους πόρους, στα δικαιώματα και στις ευκαιρίες. Έτσι θα έπρεπε να δούμε την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Βεβαίως από την άλλη, από τη μία πλευρά έχουμε τα όρια και τους περιορισμούς ε, του χάρτη και από την άλλη την, το καθεστώς της ευρωπαϊκής ηθαγένειας. Ε, ε, και τα όρια αυτά δεν είναι απόλυτα σαφή. Θα πρέπει όμως να δημιουργήσουμε αυτές τις θεσμικές προϋποθέσεις οι οποίες θα οδηγήσουν στην καλύτερη και με πιο ανθρώπινες συνθήκες διαβίωση. Ποια μπορεί να είναι στο μέλλον η σχέση ανάμεσα στον, στην Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και την ε, την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει ε, να ε, προχωρήσει αυτή η Ένωση με πιο συστηματικό τρόπο ε, έτσι ώστε να βρούμε ένα τρόπο να προωθήσουμε την συμβίωση και την άνθηση της πραγματικά ανθρώπινης ζωής. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Παλάς Τάνοκ από το Καθολικό Πανεπιστήμιο Πάσμανι Πέτερ της Βουδαπέστης. Ο κύριος Τάρνοκ συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, σε μια πρωτοβουλία δική τους και θα μας την παρουσιάσει. Ευχαριστώ. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου ε, να απευθύνω το λόγο στην Επιτροπή Λίμπε. Στην ε, παρουσίασή μου θα ήθελα να εστιάσω σε τρία βασικά σημεία σε σχέση με την ε, περσινή πρωτοβουλία για την προστασία των ε, εθνικών μειονοτήτων και τη γλωσσική επικοινομορφία. Το δεύτερο είναι η αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών και το τρίτο είναι η ενημέρωση των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα που έχουν. Καταρχάς, να αναφερθώ σε εθνοτικές μειονότητες και τη γλωσσική ποικιλομορφία. Ε, η περσινή έκθεση αναφέρει ότι οι παραδοσιακές μειονότητες είναι εκείνες οι οποίες έχουν συνυπάρξει επί σειρά αιώνων με ε, τις ε, πλειονότητες ε, Ορίζεται δηλαδή τι εστί ε, παραδοσιακή μειονότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για τα ευρωπαϊκά θεσμικά ε, όργανα να διδραματίσουν ένα ρόλο πιο ενεργό στην προστασία των μειονοτήτων. Τονίζει λοιπόν έκθεση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει ψηλά πρότυπα για την προστασία των μειονοτήτων. Η ίδια έκθεση αναφέρει τη συμφωνία πλαίσιο, τη σύμβαση πλαίσιο καλύτερα για την προστασία εθνικών μειονοτήτων και ε, τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες. Αυτά είναι κείμενα επίσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης και ε, θα ρίνει όλα τα κράτη-μέλη έκθεση, ε, τα κράτη-μέλη να κυρώσουν αυτές τις συμβάσεις και να προωθήσουν τη γλωσσική ποικιλομορφία. Όταν γίνεται λόγος λοιπόν στην Ευρώπη για την προστασία εθνικών μειονοτήτων Καταρχάς θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, εδράζεται ακριβώς και έχει ιδρυθεί ε, με γνώμονα το σεβασμό και των εθνικών μειονοτήτων. Εδώ υπάρχει πρόβλημα όμως ότι δεν υπάρχει ένα σύστημα ε, προστασίας και ελέγχου των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Τα κράτη-μέλη γενικότερα δεν θέλουν να διευρύνουν το πεδίο αρμοδιοτήτων και εξουσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ. Υπάρχουν όμως ιδιαιτερότητες και θα πρέπει να προστατεύονται ε, αυτές για να ε, διασφαλίσουμε την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Κάποιες λύσεις έχουν βρεθεί ε, τις περασμένες δεκαετίες για αυτό το πρόβλημα που είναι αρκετά περίπλοκο. Μία από τις πιο δημοφιλείς λύσεις ήταν η μεταφορά των ε, κειμένο του Συμβουλίου της Ευρώπης σε ευρωπαϊκό δίκαιο. Δεν χρειάζεται να ξαναφεύρουμε τώρα το ζεστό νερό ή το τροχό. Ε, υπάρχουν κείμενα ε, πολύ καλά και μπορούν πολύ εύκολα να ενταχθούν στο διεθνές δίκαιο και στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Η μεταφορά τους λοιπόν στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να είναι μια καλή λύση. Σύμφωνα με όλα αυτά, Πρέπει να σας αναφέρω και τις πιο πρόσφατες επιτυχίες. Μια επιτυχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο ενέκρινε ψήφισμα στις 7 Φεβρουαρίου ενιστότους έτους, το οποίο αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρει ευθύνη για την προστασία και πρόθεση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και θεωρεί απαραίτητο να βελτιωθεί το νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να προστατεύονται και να διαφυλάσσουν τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες. Το ίδιο ψήφισμα τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στερείται αποτελεσματικών εργαλείων για να παρακολουθεί και να ελέγχει το σεβασμό των ε, μειονοτικών δικαιωμάτων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το τονίσουμε, διότι η παρακολούθηση και ο έλεγχος είναι κάτι κρίσιμο πάντα. Το ίδιο ψήφισμα ζητεί αποτελεσματική ε, παρακολούθηση και έλεγχο της κατάστασης παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτοχθόνων και γλωσσικών μειονοτήτων. Άλλο σημείο κλειδί που τονίζει ότι η προστασία των μειονοτήτων είναι πολύ σημαντική. Αυτόχθονες και γλωσσικές μειονότητες ηθαγενείς, που ποτέ δεν έχει αναφερθεί σε τέτοιο ψήφισμα με τέτοιο τρόπο αυτό. Δεύτερο, η ε, μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Πολιτών. Υπάρχει μια σχετική έκθεση που καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθεωρήσει ε, τις ε, διαδικασίες, το παραδεκτό, διαδικασία ε, καταχώρησης μιας τέτοιας πρωτοβουλίας και μια ε, νομική γνωμοδότηση που συνάπτεται τονίζει ότι υπάρχουν ε, γενή προβλήματα και δυσλειτουργίες που πρέπει να διορθωθούν στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών. Ε, Ξέρουμε τι γίνεται στην πραγματικότητα. Από το 2012 στην καθημερινή ζωή με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών ακούμε πολλά επιχειρήματα ότι χρειάζεται αναθεώρηση και βελτίωση αυτή η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία. Μετά την πρώτη τριετία που έγινε μια αξιολόγηση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε μια έκθεση για την πρωτοβουλία αυτή το 2015, τον Οκτώβριο συγκεκριμένα. Ε, και στο προηγουμένως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης εξέδωσε αντίστοιχη πρόταση και έκθεση χωρίς να εντοπίζει ότι υπάρχουν. Ε, ο Φρανς Τίμερμανς ε, ανακοίνωσε σε μια σχετική ημερίδα επιτέλους ότι θα προβεί σε αναθεώρηση της πρωτοβουλίας αυτής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τώρα την Τετάρτη ας πούμε ε, στις Επιτροπές ΑΦΚΟ και ΠΕΤΗ θα υπάρξει δημόσια ακρόαση για να αναθεωρηθεί το νομικό ότι υπάρχει ε, αυτό το εργαλείο και επίσης είναι πολύ τε εγκρίνει μάλλον ένα σχέδιο ε, εκστρατείας ενημέρωσης στα θα έρθουν πιο κοντά οι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα ε, θα συμμετέχουν περισσότερο και στις ευρωεκλογές όπου η αποχή ήταν τεράστια πρωτοβουλία για την προστασία των μειονοτήτων και εγώ συμμετέχω στην Ουγγαρία στη σχετική πρωτοβουλία. Όπως είδαμε τους τελευταίους μήνες υπάρχουν τεράστια προευρωπαϊκή ηθαγένεια ιδιαίτερα ως προς το ποιο είναι τα δημοκρατικά εργαλεία που διαθέτει ο πολίτης και που είναι άγνωστα στην ε, Ένωμη Πολιτών. Έτσι λοιπόν, αν δεν μπορούμε να ενημερώσουμε τους πολίτες για τα δικαιώματά τους, χάνουμε το στόχο γενικότερα και της Ευρωπαϊκής προσώπων που ανήκουν σε εθνοτικές και γλωσσικές μειονότητες και να ενισχύσει ε, την ποικιλομορφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολιτισμική και γλωσσική εξ προθεσμία λέγει στις 3 Απριλίου. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 600.000, 650.000 μάλιστα ε, υπογραφές ε, πανευρωπαϊκά. Κάποια γλωσσική αυτόχθονη παραδοσιακή μειονότητα στην Ευρώπη. Είναι δύσκολο να κινητοποιηθούν αυτές οι κοινότητε και τα πρόσωπα που ανήκουν σε αυτές. Οι συλλογές στα δικαιώματά του. Αυτό θα πρέπει να βελτιωθεί. Και τέλος κάτι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου. Αν και υπήρξαν επιτυχίες, όπως το έδειξε το πρόσφατο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τζίλιαν Μουρ, που ε, προσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα μας δώσει ε, την άποψη Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε κάποια από αυτά τα ε, θέματα και τις πτυχές αυτές. Έχετε το λόγο. Thank Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα αναφερθώ στην έκθεση της Επιτροπής για την ιδιότητα του πολίτη, την Ευρωπαϊκή Υπηκότητα. Δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 24 Ιανουαρίου του 2017. Τι περιλαμβάνει. Είναι ένα έγγραφο στραμμένο καταρχάς στο μέλλον. Δίνει την δυνατότητα να δούμε το τι μπορεί να κάνει καλύτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ενισχύσει τα δικαιώματα των πολιτών. Είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία. Δημοσιεύθηκε μαζί με την έκθεση για το άρθρο 25 που είναι μια πιο τεχνική έκθεση που απαιτείται από τη συνθήκη. Ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες στην εφαρμογή συγκεκριμένων δικαιωμάτων των πολιτών. Πώς εμείς λοιπόν συνδυάζουμε τις δύο αυτές εκθέσεις. Η κυρία Κωνστακοπούλου αναφέρθηκε στην πολυεπίπεδη πολιτική που ακολουθείται, σχεδιάζεται και ακολουθείτε. Αυτό ισχύει για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο εσωτερικό των ε, εσωτερικών ε, τμήματων και διευθύνσεων συνεργαζόμαστε με οριζόντιο τρόπο, δεν περιοριζόμαστε δηλαδή ε, ο καθένας στο τμήμα του, φυσικά συνεργαζόμαστε και με το κοινό μέσο διαβουλεύσεων, λαμβάνουμε υπόψη το ευρωμαρόμετρο, και τον Μάρτιο του 16 ίσως να ε, θυμίστε ότι είχαμε μια κοινή ακρόαση με την ε, Επιτροπή σας, με την Πέτη και την Τζούρι ε, σχετικά με το θέμα της ευρωπαϊκής υπηκότητας. Νομίζω ότι αυτά έδωσε, αυτό έδωσε πολλά καλά στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις εκθέσεις που ακολούθησαν. Εμείς δημοσιεύουμε λοιπόν την έκθεση αυτή και τι συμβαίνει μετά. Υπάρχει μια διαδικασία θεσμικής επεξεργασίας των επιτελεσμάτων αυτών των εκθέσεων και μετά από τη δημοσίευση πέρυσι το Συμβούλιο ε, υιοθέτησε τα δικά του συμπεράσματα ε, ε, πέρυσι. Έγινε συζήτηση επίσης στις αρχές Δεκεμβρίου και στην Επιτροπή των Περιφερειών και τελικά το Κοινοβούλιο υιοθέτησε την έκθεση για την Ευρωπαϊκή Υπηκότητα την 12η Δεκεμβρίου του 2017. Υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία λοιπόν που ακολούθησε τη δημοσίευση της έκθεσης. Σας ευχαριστούμε για τη συνέχεια που δώσατε. Ιδιαίτερα η έκθεσή σας ε, περιλαμβάνει πάρα πολλά θέματα στα οποία ζητάτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει ε, προσεκτικά. Τώρα για την ίδια την έκθεση διαφρώνεται γύρω από τέσσερις βασικές προτεραιότητες ή θεματολογίες. Εγώ θα σας παρουσιάσω τις θεματολογίες αυτές και θα αναφερθώ σύντομα σε ε, το τι κάνουμε γύρω από αυτά. Το πρώτο θέμα είναι η, προμό, η προώθηση ε, των κοινών αξιών και δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την έρευνα την οποία κάναμε, ιδιαίτερα το Ευρωβαρόμετρο μας δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι συνειδητοποιούν την ιδιότητα αυτή, αλλά θέλουν να γνωρίζουν περισσότερα για τα δικαιώματά τους. Δεν τα γνωρίζουν όλα. Το μας δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι συνειδητοποιούν την ιδιότητα αυτή, αλλά θέλουν να γνωρίζουν περισσότερα για τα δικαιώματά τους. Δεν τα γνωρίζουν όλα. Κρατία ενημέρωσης και συνειδητοποίησης των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών. Ελπίζω να δείτε τους καρπούς της εκστρατείας αυτής να παίρνουν ε, πολιτών για το δικαίωμά τους σε επίπεδο προξενικής προστασίας, αν έχουν ανάγκη ας πούμε προστασία σε μια τρίτη χώρα είναι ένα δικαίωμα το οποίο λίγοι γνωρίζουν, η λεγόμενη προξενική προστασία εταίρου. Ε, και όταν κάποιος μένει νόμιμα σε μια τρίτη χώρα, σε μια άλλη χώρα μέλος. Στα πλαίσια της προώθησης λοιπόν των κοινών δικαιωμάτων και των κοινών αξιών και στα πλαίσια της προστασία των δικαιωμάτων εμείς φέτος θα κυκλοφορήσουμε εμείς συγκρίνουμε τις νομικές ρυθμίσεις και αξιολογούμε τα αποτελέσματα. Ένα δεύτερο σημείο είναι στην έκθεσή μας η προώθηση της βελτίωσης της συμμετοχής των πολιτών στην δημοκρατική ζωή της Ευρωπαϊκής Ζωής της Ένωσης. Ένας κλάδος αυτής της, της κατάστασης είναι αυτό το οποίο ήδη προανέφερα, δηλαδή ανάγκη για μεγαλύτερη ενημέρωση, πληροφόρηση, συνειδητοποίηση των δικαιωμάτων συμμετοχής στις εκλογές, η συλλέξη της βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την δυνατότητα συμμετοχής στις εκλογές, έτσι ώστε οι πολίτες να μην χάνουν το δικαίωμα ψήφου όταν μετακινούνται σε άλλη πόλη και χώρα. Φέτος οργανώνουμε και μια τεχνική συνάντηση για να βελτιώσουμε το ποσοστό συμμετοχής των Ευρωπαίων σε δημοτικές εκλογές σε άλλες χώρες. Προστασία λοιπόν της συμμετοχής σε δημοκρατικές διαδικασίες για την αύξηση του ποσοστού των νέων και των ευάλωτων κατηγοριών όπως οι γυναίκες και οι ανάπηροι η έκθεση να κάνει είναι να δει τι γίνεται με τη γραφειοκρατία, να καταστήσει πιο εύκολες τις μετακινήσεις των πολιτών από χώρα σε χώρα, να καταστήσει απλούστερες τις διοικητικές διαδικασίες που ε, δημιουργούνται όταν ε, πηγαίνει. Δηλαδή η βασική ιδέα είναι να επιτρέψουμε στον πολίτη να ολοκληρώνει online επιγραμμικά τις υποχρεώσεις του και τις δικηστικές διαδικασίες και θα προτείνουμε ένα προσάρτημα συγκεκριμένων ε, διαδικασιών για θέματα όπως της ασφάλειας και η προώθηση της ισότητας είναι ένα διτό θα έλεγα θέμα. Εδώ έχει ξεκινήσει πολλή δουλειά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διάφορα τμήματα αυτού του, αυτού του θέματος. Προώθηση λοιπόν της ισότητας, η Ευρωπαϊκή Επιρρηνούπολης για την καταπολέμηση της βίας και η οδηγία για την ισορροπία επαγγελματικής σταδιοδρομίας και προσωπικής ζωής για τα θέματα της ασφάλειας, το Ευρωβαρόμετρο δείχνει ότι ανησυχούν οι πολίτες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται τη ζωής για τα θέματα της ασφάλειας, το Ευρωβαρόμετρο δείχνει ότι ανησυχούν οι πολίτες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται στα πλαίσια ενός σχεδίου για ενιαίες εθνικές ταυτότητες και αποδεικτικά έγγραφα ε, έτσι θα βελτιωθεί το αποδεκτό και η επαλήθευση και ο έλεγχος των εγγράφων αυτών και θα διευκολυνθεί η καθημερινότητα, αλλά ταυτόχρονα και παράλληλα με όλα αυτά, εμείς προσπαθούμε να δούμε πώς θα βελτιώσουμε και θα ενισχύσουμε την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη, για το πώς θα ενισχύσουμε την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη και ελπίζω να μπορέσω να ενημερώσω την ομάδα αυτή και για τη σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Ε, όλη τη... Η κυρία Σπινέλη, Κόμες, Έγκελ, Τσάκη και η Σοφή Νετφέλτς. Η κυρία Σπινέλη πρώτη, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα ιδιαίτερος να ευχαριστήσω του. Θα υποβάλω συνθετικά. Η πρώτη αφορά τον ε, καθηγητή κύριο Κόσενοφ ε, κοσμοπολίτικου ας πούμε νόμου ε, από ε, άλλες ε, πιο παραδοσιακές αρχές. Δεν είναι αυτή η ιδέα του Φερχότσταρτ. Η ιδέα ακριβώς του κράτους δικαίου και της δικαιοσύνης για όλους. Το δεύτερο, όταν λέτε ότι η ιδέα της των βασικών αρχών ας πούμε της ε, ε, ιδέας και το, της αρχής ε, των δικαιωμάτων των πολιτών λοιπά Δεν νομίζω ότι το άρθρο 50 προκαλεί κάποιο πρόβλημα σε αυτά τα δικαιώματα, αλλά η ιδέα της διατήρησης της ευρωπαϊκής ηθαγένειας για αυτούς τους πολίτες έχει σαν σκεπτικό, σκεπτικό το γεγονός ε, ότι θα πρέπει να έχει κανείς τη δυνατότητα να κάνει τις ε, επιλογές στη ζωή του βασιζόμενος ε, στις δυνατότητες που του παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Αυτή η εγγύηση τους δόθηκε με, τρόπο μόνιμο για όλη τους τη, ε, τη ζωή. Ε, επομένως κάτι θα πρέπει να γίνει. Ε, λέμε ότι οι ε, Βρετανοί πολίτες ψήφισαν για να χάσουν δικαιώματα και αυτό είναι το επικίνδυνο, η επικίνδυνη σκέψη της κυβέρνησης της, του Ηνωμένου Πολιτείου. Θα ήθελα να, να κάνω και κάποια ερώτηση στην κυρία Τζίλιαν Μόρ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν ε, κάνει λόγο ε, στα, ε, στην διασφάλιση της ασφάλειας μέσα από δυνατότητες που έχουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην κυρία Ντόρα Κωστακοπούλου, την καθηγήτρια Ευρωπαϊκού Δικαίου, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αναφέρεστε σε κοινωνικά δικαιώματα. Θεωρείτε χρήσιμη ε, την ε, αποδοχή της, Ευρωπαϊκής, της ε, Χάρτας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτήν, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στον 10 καθηγητή Τάρνοκ, ο οποίος αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία των Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία, αυτή η ECI πραγματικά είναι θρησιγενής. Πνέει τα λίστια, το γνωρίζουμε γιατί δεν δόθηκε ποτέ καμία συνέχεια σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία. Και σας ρωτώ λοιπόν το εξής, πώς είναι δυνατόν και μέσα από τις τροποποιήσεις που θα γίνουν στην πρόταση της Κομισιόν, πώς είναι δυνατόν να ενταχθούν ε, οι αιτιολογήσεις ε, του ε, Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και όσον αφορά το TPIP και το ΣΕΚΑΤ το Safe Pack μάλλον. Το Safe Pack είναι η δυνατότητα ε, ε, ε, μερικής καταγραφής των πρωτοβουλειών και το άλλο αφορά στη δυνατότητα επανορισμού της έννοιας του Legal Act. Και εδώ η Κομισιόν καλείται να υποβάλει προτάσεις τροποποίησης ε, μετά από μια επιτυχή πρωτοβουλία των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Δεν πρόκειται αυτό να αφισβητήσει το άρθρο 50. Η καθηγήτρια κυρία Κωνστακοπούλου, για αυτή την έννοια του πολιτισμού, ότι είναι ο εξανθρωπισμός του ανθρώπου στην κοινωνία. Τα ε, προγράμματα για τις χρυσές θεωρήσεις διαβατηρίων ή τα επενδυτικά, όπου τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολλούν και με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται το ξέπλυμα του χρήματος και η εισαγωγή του εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς το βλέπετε αυτό. δεν ε, θα πρέπει να τους προσφορά προς μια χώρα. Εδώ μιλάμε για οργανωμένη πώληση ευρωπαϊκής ηθαγένειας. Γι' αυτό το έχουν στήσει τα κράτη-μέλη τα ίδια. Πώς σκέφτηκε η Επίτροπος κυρία Γιούροβα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο κύριος Στίμερ μας δεν το καταλαβαίνει αυτό, δεν αναλαμβάνεται. Θα ήθελα την άποψή σας παρακαλώ, Ζωβάνε και ζητώ συγγνώμη για τη φωνή μου. Την περασμένη εβδομάδα ήμουν στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και κρυολόγησα. Λοιπόν, ε, στη φωνή έχω πρόβλημα, όχι ε, στη σκέψη. Ε, θέλω να σας υποβάλω λοιπόν μερικά σημεία για να τα μοιραστώ μαζί σας. Πρώτον, περιέργως, και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η ακρόαση αυτή ανάγεται σε μια παλιά δική μου πρωτοβουλία. Γιατί ήθελα να ακούσω και από εσά και από άλλους που δεν έχουμε καλέσει, αλλά δεν βρίσκω και κανένα δύσκολο να βρει ε, δημοσιεύματα σχετικά. Πώς θα μπορούσαμε να προωθήσουμε την αρχή της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας που κυκλοφορεί από την εποχή της συνθήκης και αυτό δεν το έχω ακούσει. Πώς θα τη μεταξελίξουμε. Ε, πέρα από κάποια ακαδημαϊκά και πολύ άσχετα πράγματα. Περί τίνος πρόκειται στην Ιθαγένεια. Τι είναι η Ιθαγένεια στον 21ο αιώνα σε μια τέτοια κοινωνία. Από κάποια ακαδημαϊκά και πολύ άσχετα πράγματα. Περί τίνος πρόκειται στην Ιθαγένεια Τι είναι η Ιθαγένεια στον 21ο αιώνα σε μια τέτοια κοινωνία. Και αυτό ίσχυε και για την δεκαετία, την τελευταία τουλάχιστον του 2000 που υπεγράφει η συνθήκη του Μαστρίχτ. Είναι Ευρωπαίος πολίτης με γεια σου με χαρά σου αφού αποφάσισε ότι δεν σου λέει τίποτα Ευρωπαϊκή Ένωση στο καλό. Κανένας Βρετανός πολίτης που θα... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ και τους τρεις εκπροσώπους του ακαδημαϊκού κόσμου. Ήρθα λίγο αργότερα και δεν άκουσα ε, τα πάντα. Όταν μιλάμε για ευρωπαϊκή Ιθαγένεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εκτός αυτής ε, φαίνεται ότι γίνεται όλο και περισσότερο κάτι που αποκλείει και δεν συμπεριλαμβάνει ε, κάτι που μας διαχωρίζει από τους άλλους και μας κάνει απόμακρους. Δύο θέματα πρέπει να αναφερθούν. Ε, και πραγματικά ε, εντυπωσιάστηκα από τα όσα είπε ο Ρέφος Έγγελ. Το θέμα των χρυσών βίζων και το θέμα των golden visas ε, και το θέμα του Brexit. Ξέρω ότι και για τα δύο πράγματα έχεις διαφορετική προσέγγιση γιατί μπορώ να συμφωνήσω με αυτά που είπες για αυτή τη διαδικασία που δίνονται οι χρυσές βίζες. Δεν είναι γιατί κάποιος έγινε καλό μέλος, απέδειξε ότι είναι καλό μέλος της κοινότητας αλλά γιατί έχει διοχετεύσει χρήματα στην ιδιωτική αγορά. Ε, επομένως, ναι, το θέμα αυτό ε, καλά το ανέφερε ο, ο Φρανκ, ότι θα πρέπει οπωσδήποτε οι άνθρωποι αυτοί να ταυτίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μετά ε, μας τα χάλασε με το Brexit ε, γιατί, και τις παρατηρήσεις του, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επειδή κάποιοι άλλοι ψήφισαν με συγκεκριμένο τρόπο θα απεκδηθούν των δικαιωμάτων τους που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Μα οι ίδιοι πρότειναν ε, να πληρώσουν και κάποια χρήματα, λίγα, ε, έτσι ώστε να διατηρήσουν την ε, ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Αυτό από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά διατηρούμε αυτό το σύστημα της χρυσή βίζας. Επίσης, ε, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια υπόθεση ενώπιον των ε, ε, Ολλανδικών δικαστηρίων. Ένας Βρετανός υπήκος που ζει στην Ολλανδία ζήτησε από το δικαστήριο να μελετήσει εάν αυτομάτως το Brexit σημαίνει και κατάργηση της ευρωπαϊκής ηθαγένειας γιατί η ευρωπαϊκή ηθαγένεια είναι συνδεδεμένη με την εθνική αλλά είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Δύο ερωτήσεις. Ε, πρώτον, θα ήθελα και οι τρεις σας ε, να μου πείτε ε, την άποψή σας για τον Bill of Rights. Δεύτερον, κυρία Μόρ, ως εκπρόσωπο της Κομισιόν, άκουσα αυτό που είπατε για την εναρμόνιση των ταυτοτήτων και μου σηκώνεται λίγο η τρίχα και λέτε για λόγους ασφαλείας. Εγώ το βλέπω σαν ένα επιπλέον μέτρο ασφάλειας που το βάζουμε από την πίσω πόρτα και που θα έχει επίδραση στην ε, ε, ηθαγένεια. Και επίσης, απλά για να καταγραφεί, το θέμα της πρωτοβουλία, Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας ε, Πολιτών εγώ νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι θεσμοί της να γίνουν πολύ πιο δημοκρατικοί και να αφήσουμε αυτά τα παιχνιδάκια ε, που δίνονται κάθε τόσο. Γιατί φαίνεται ότι μιλάμε για κάποιες πρωτοβουλίες τις οποίες θέλουμε να δώσουμε περισσότερο βάρος από ότι ε, τα ε, εκατομμύρια πολιτών που ψήφισαν στις τελευταίες ευρωπαϊκές εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που φαίνεται να το ξεχνά. Ευχαριστώ. Κυρία Σέπελ, ευχαριστώ Πρόεδρε Μειονοτήτων. Και εδώ πάλι είμαι σε κάποια σύγχυση. Γιατί όλοι οι πολίτες μας θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα, άνδρες και γυναίκες. Ακόμα πλήρωναν τους πολίτες για τα δικά τους δικαιώματα ως πολίτες των εθνικών κρατών. Γιατί από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσουμε και εκεί είναι το πρώτο μεγάλο έλλειμμα. Και αν έκαναν ταινία, ακόμα και οι εθνικοί. δεν θα πρέπει να πωλείται. Να υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αλλά οι κανόνες διαφέρουν στις περιπτώσεις διαφθοράς, άρα το θεωρώ κάπως ανάρμοστο αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ θέσεις ε, που έπρεπε να δουλέψω ήταν ακριβώς αυτό της ε, ηθαγένειας. Ε, μεταρρύθμιση της ηθαγένειας έτσι ώστε να ξεκινήσουμε επί τη διαδρομή που διανύουν και πολιτιστική διαδρομή που διανύουν τα νέα παιδιά τα οποία έρχονται στην χώρα. Και επομένως να έχουμε μια κανονική διασύνδεση ανάμεσα στην Ιταλία. Με τελείως διαφορετικό τρόπο δηλαδή μπορεί να επιτύχει την υπηκότητα κάποιος στις χώρες. Και επομένως το πρώτο βήμα θα πρέπει να είναι κάποια σύνδεση ανάμεσα στην υπηκότητα του κράτου μέλους με την ε, ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Γιατί μερικοί λένε δεν υπάρχει λόγο να γίνει τώρα η μεταρρύθμιση. Θα πρέπει πρώτα η Ευρωπαϊκή Ένωση να δουλέψει πάνω στο να τροποποιήσουν τι αρχέ που διέπουν την εθνική ηθαγένεια. Ε, γιατί πέρα από το ότι δεν αναγνωρίζουν ε, πολύ ότι τα παιδιά τα οποία γεννιούνται και μεγαλώνουν σε υπηκότητα. υπηκότητας. Ευχαριστώ. Η Εγώ για τους κοφούς ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εθνικές υπηκότητες, ηθαγένειες στα κράτη-μέλη. Αλλά οι κοφοί πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουν μεγάλα εμπόδια, πρόσβαση στην επικοινωνία και στην ενημέρωση γιατί δεν ακούν. Όταν μιλούμε λοιπόν για την προώθηση ε, της κουλτούρας της νοηματικής γλώσσας, γιατί συχνά τους λησμονούμε. Μιλάμε συχνά για τις ομιλούσες γλώσσες, αλλά όχι για την νοηματική. Πώς θα συμπεριληφθούν λοιπόν οι κοφοί σε αυτή την έννοια της ε, γλωσσικής επικοινομορφίας και πώς θα γλώσσες. Αυτοί μπορούν να θεωρηθούν γλωσσική μειονότητα. Κατά την άποψή μου, ναι. Εγώ αυτό πιστεύω. Εγώ θεωρώ ότι ανήκω σε γλωσσική μειονότητα. Θα ήθελα κι εσείς να μου το επιβεβαιώσετε, αν υπάρχει αυτό στο πλαίσιο αναφοράς ε, για τους κοφούς πολίτες ε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω. Με ευρύτατη πλειοψηφία το Κοινοβούλιο. Και θα ήθελα να μάθω πραγματικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν προτίθεται να δώσει κάποια συνέχεια και ποια στο ψήφισμα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως και άλλα θεσμικά όργανα ευρωπαϊκά να παίξουν το ρόλο που τους αναλογεί και για την νοηματική και για τους χρήστες της νοηματικής. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχει ζητήσει το λόγο κανείς άλλος συνάδελφος. Πολύ ενδιαφέροντα τα σημεία που τέθησαν. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στους ομιλητές μας για να απαντήσουν. Ο καθηγητής Κουτσενόφ. Με την ίδια σειρά. Όπως και προηγουμένως. Σας ευχαριστώ για τις εξαιρετικές σας ερωτήσεις. Υπάρχει ένα κοινό επίπεδο κατανόησης θα έλεγα, μπορούμε να βασιζόμεθα σε αυτό. Θα ήθελα καταρχάς ξεκινώντας να αναφερθώ στα του Brexit. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Έγγελ, όχι όμως ε, για τον λόγο γιατί ψήφισαν να φύγουν, αλλά γιατί το άρθρο 50 το οποίο είναι σε αντίθεση με τη ρύθμιση της συνθήκης που λέει ότι οι συνθήκες έχουν αόριστη διάρκεια. Εδώ προφανώς υπάρχει ένα όριο. Εγώ δεν θέλω τώρα να φανώ νομικιστής, αλλά το 50 προϋποθέτει την δυνατότητα αποχώρησης. Ο πρώτος πυλώνας λοιπόν είναι η εσωτερική αγορά και ο δεύτερος πυλώνας είναι η ιδιότητα του πολίτη. Αν βασιστούμε λοιπόν στη συνθήκη δεν είναι δυνατόν να διαφυλάξουμε, ε, αν βασιστούμε λοιπόν στη συνθήκη δεν είναι δυνατόν να διαφυλάξουμε ε, τερμηνίες τότε θα αντικαταστήσουμε την άποψη των Άγγλων με τη δική μας άποψη και θα αντικαταστήσουμε τελικά και την άποψη εμείς να αγνοούμε τις δημοκρατικές εξελίξεις οι οποίες στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μας αρέσουν. Το θέμα είναι ότι στον κόσμο που επιτρέπει να γίνεται διάκριση ανάμεσα σε πολίτες και μη πολίτες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, αυτό το ονομές πολίτες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένας μη πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έφτασε στο Λουξεμβούργο, στην που έχουμε δημιουργήσει και εκτός των δικαιωμάτων που έχουμε δημιουργήσει, όλους τους πολίτες τρίτων χωρών που δεν έχουν την υπηκαότητα. Αυτό εγώ δεν εκπροσωπώ την κυβέρνηση της Μάλτα, δεν είμαι ε, από τη Μάλτα. Εγώ συνεργάζομαι με τις αρχές της Μάλτα. να δούμε με μεγάλη ψυχραιμία. Νομίζω ότι υποδειγματικά μας παρουσιάζει την προστιθέμενη αξία της Ένωσης που δημιουργήσαμε. Ο ακριβώς αυτό. Ένας πολίτης στο Ταλίνα και ένας πολίτης στο Λουξεμβούργο πρέπει να έχει τα ίδια δικαιώματα με μια Ιταλίδα ή ο κόσμο γεννιέται με ένα συγκεκριμένο καθεστώς. Δεν επιλέγεται αυτό λόγο θρησκείας ή λόγω αξιών ή λόγω προσδοκίων. Ξέρω ότι δεν είναι πολύ δημοφιλές αυτό που λέω. Είναι ότι δεν υπάρχει καμία δεοντολογική ή ηθική διάσταση στο εσωτερικό. Ας φανταστούμε ότι ο κύριος Σέγγελ είναι φιλοαμερικανός. Πηγαίνει αύριο στις Ηνωμένε Πολιτείες με το διαβατήριο. Το Ρωμά. Ε, αυτό συνεργάζεται με δομές των κρατών μελών και φόρα και προφανώς ε, το καλωσορίζουμε. Η Ιθαγένεια. Ε, Σας ευχαριστώ. Τέθηκε ένα ερώτημα για την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ε, έγγραφα των παραμενόντων σε μια χώρα και για τα δελτία ταυτότητας. Προβλέπεται λοιπόν μια ανακοίνωση το 18, προετοιμάζουμε μια μελέτη επιπτώσεων και νομίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί στις 17 Απριλίου. Υπάρχουν δύο τμήματα. Καταρχάς οι κάρτες παραμονής από τη μία και οι ταυτότητες από την άλλη. Τα έγγραφα παραμονής σύμφωνα με το θέμα όπως τίθεται τώρα καλύπτει τα μέλη της οικογένειας. Υπάρχουν ας πούμε άνθρωποι σαν και εμένα οποίοι ζουν στο Βέλγιο. Δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο έγγραφο ειδικό για μένα. Μπορεί να πάρω μια ταυτότητα παραμονής για ξένους και αυτό δημιουργεί σύγχυση σε άλλες χώρες. Είναι ένα απλό έγγραφο και αυτό το οποίο εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της μελέτης επιπτώσεων είναι να δούμε αν υπάρχει κάποιος τρόπος Να υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα να ισχύουν ενιαία στοιχεία στις περισσότερες ε, κάρτες παραμονής. Και λέω εδώ στην κυρία Σπινέλη ότι αυτό δεν έχει σχέση με το ειδικό καθεστώς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα άλλο τμήμα των πρωτοβουλειών μας είναι οι κάρτες, τα δελτία ταυτότητας. Η ε, οδηγία για την ελεύθερη διακίνηση σας δίνει τη δυνατότητα να μετακινήσετε ελεύθερα και σε εξωτερικό σύνορο με ταυτότητα ή με διαβατήριο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο λοιπόν και λόγω της σημασίας που έχει η κάρτα ταυτότητα σε θέματα ασφαλείας το πρέπει να μας πιέσει να καταλάβουμε ακριβώς τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει αν οι κάρτες που κυκλοφορούν είναι λειτουργικές. Βασική ιδέα είναι λοιπόν να διευκολύνουμε την ελεύθερη διακίνηση, να βελτιώσουμε την ασφάλεια. Δεν θέλουμε να εναρμονίσουμε τις εθνικές ταυτότητες. Κάθε χώρα έχει τα δικά της, κάποιες χώρες χρησιμοποιείται με διαφορετικό τρόπο. Στο Βέλγιο το χρησιμοποιούμε όταν πηγαίνουμε στο φαρμακείο ας πούμε. Πάντως ε, είναι σαφές να υπάρχουν κάποια δεδομένα επίπεδα ασφαλείας στις κάρτες αυτές. Πάντως δεν έχουμε εντοπίσει ακόμα τις σωστές επιλογές και τις προτάσεις που θα κάνουμε. Η μελέτη συνεχίζεται. Το δεύτερο θέμα έχει σχέση με την ανάγκη εναρμόνισης της διαδικασίας απόκτησης υπηκότητας. Πολλοί είπαν ότι στα πλαίσια του ευρωπαϊκού δικαίου η υπηκότητα εντάσσεται στις αρμοδιότητες των κρατών μελών στο βαθμό που το κράτος μέλος δίδει ή αποσύρει την υπηκότητα με βάση τον κοινοτικό νόμο. Εδώ τίθεται το θέμα και σε σχέση με τις δυνατότητες απόκτησης εγγράφων μέσω επενδύσεων και έχει αναφερθεί και η Επιτροπός Γιουρόβα ότι πριν το τέλος του χρόνου η Επιτροπή θα δημοσιεύσει μια έκθεση για τα εθνικά προγράμματα χορήγησης υπηκότητας στους επενδυτές. Εμείς συνεχίζουμε τις μελέτες τώρα, βλέπουμε τι ισχύει σε κάθε χώρα βλέπουμε τι ισχύει στις εθνικές νομοθεσίες, βλέπουμε ποιες είναι οι κατευθυντήριες γραμμές και ελπίζουμε πριν το τέλος του χρόνου να μπορέσουμε να δημοσιεύσουμε μία σειρά προτάσεων. Ένα τρίτο σημείο είναι αυτό που έθεσε η κυρία Στίβενς για την ειδική γλώσσα των κοφαλάλων. Δεν μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένες απαντήσεις εδώ, αλλά όπως έχω ήδη πει, Έχουμε μια ομάδα εργασίας για την υπηκότητα, συνεργαζόμαστε και με άλλα τμήματα της Επιτροπής και γνωρίζω ότι συνεργάζονται ε, για να βελτιώσουν την πράξη για την προσβασιμότητα, όπως επίσης και την επικύρωση της σύμφασης του Μαρακές. Και ε, συγκρατώ αυτό το οποίο είπε σχετικά με τα θέματα που παραμένουν ανοιχτά. Θα οργανώσουμε αυτή τη συνάντηση πριν το τέλος του χρόνου για την ε, μεγαλύτερη συμμετοχή στις δημοκρατίες. ...του Κοινοβουλίου, οπότε δύσκολο να ε, βρεθεί κάποια συμφωνία. Αυτά. Σε γενικές γραμμές έχω να πω μέχρι στιγμής. Ευχαριστώ πολύ Σοφή. Δεν ξέρω αν θέλει κανένας βουλευτής το λόγο. Ναι, πραγματικά έπρεπε να τα συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Χαίρομαι πάρα πολύ ε, και σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Είναι προφανές ότι ο καθένας μας έχει διαφορετικές ε, θεωρήσεις για το θέμα αυτό. Και τα διάφορα κράτη-μέλη μπορεί να διαφωνούν μεταξύ τους ε, ή να συμφωνούν και με ευρωπαϊκή σκοπιά. Ποια είναι εκείνα τα θέματα στα οποία έχετε ήδη συμφωνήσει, θα με ενδιαφέρει να μου πείτε. Πού καταφέρατε να βρείτε ε, ένα κοινό έδαφος. Πρώτα στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μετά με το Συμβούλιο. Και ποια είναι τα κύρια ζητήματα και τα κύρια προβλήματα που καλείται να λύσει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και δεν διαφωνεί με το Συμβούλιο. Η κυρία Ντφέλτ. Είναι αρκετά για να είμαι ειλικρινής. Σαφής. Εγώ διαπραγματεύομαι βάσει της εντολής που έχει εγκριθεί στο Κοινοβούλιο. έχω ένα ξεκάθαρο στόχο να είναι όσο γίνεται ευρύτερη πλειοψηφία, γιατί το θέμα είναι λεπτό και ευαίσθητο και δεν μπορεί να περάσει με ε, περιστασιακή μικρή πλειοψηφία. Χρειάζεται πλειοψηφία και στο Συμβούλιο. Εγώ μπορώ να σας ενημερώσω για τις λεπτομέρειες. Στα θέματα που έχουμε συμφωνήσει βασικά είναι λεπτομέρειες. Τα μεγάλα θέματα εκκρεμούν οι νέε διατάξεις που θέλει να εισαγαγεί το Συμβούλιο για να περιορίζει ουσιαστικά και σε μεγάλο βαθμό την κυκλοφορία τους και την ελευθερία τους, δεν είναι κράτηση αυτή καθ' αυτή, είναι περίπου κράτηση. Σε ορισμένα κράτη-μέλη, όπως η Γερμανία, όπου έχουν περιφερειακό σύστημα για την υποδοχή στα ομόσπονδα κρατήδια και βάσει της διοικητικής δομής έχει νόημα να πεις ότι δεν μπορεί κάποιος να φεύγει από ένα γεωγραφικό χώρο. Αλλά αυτό θα μπορούσε να ερμηνευθεί ε, ότι έχουν το δικαίωμα τα κράτη-μέλη να, να κλειδώνουν κάποιον, ας πούμε, σε ένα γεωγραφικό χώρο. Ότι εντάξει δεν είσαι σε κράτηση, αλλά δεν μπορείς και να κουνηθείς από εδώ. Αυτά θα πρέπει να τα λύσουμε, γιατί τα κράτη-μέλη το Συμβούλιο δεν ξεκαθαρίζει γιατί χρειάζεται αυτές τις διατάξεις. Ε, μας λένε συνεχώς ότι πρέπει να κωδικοποιήσουμε σε νόμο αυτό που ήδη κάνουμε. Μα αν το κάνουν κάτι είτε δεν χρειάζεται νομοθεσία είτε κάτι κάνουν που είναι παράνομο. Όπως και για την ενημέρωση. Εμείς θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε τι είδους πληροφόρηση θα έχουν οι άνθρωποι αυτοί. Και κατά την άποψή μας, όσο πιο ενήμεροι είναι, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να ε, δημιουργήσουν προβλήματα αργότερα. Και δεν καταλαβαίνω το Συμβούλιο γιατί θέλει να περιορίσει ε, την ενημέρωση και να μην έχουμε λίστες και να μην έχουμε ε, αιτιολογικές σκέψεις ότι θα πρέπει να τους δίνουμε ενημέρωση για αυτά και για αυτά. Διαφωνούμε επί της φιλοσοφίας. Δεν λέω ότι δεν θα συμφωνήσουμε, εύκολο πάντως δεν θα είναι. Θα κάνω ό,τι μπορώ ε, για να επιτύχω όλα αυτά που ζήτησε το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Φτάνουμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερησίας διατάξεως σχετικά με την κατάσταση των πραγμάτων καθώς επίσης και την, ε, τις διαβουλεύσεις όσον αφορά την επανεγκατάσταση του Ψηφιακού Κανονισμού 516-2014. Τρεις, ε, ε, δύο τριμερείς διάλογοι έχουν οργανωθεί, Δεκέμβριο και Ιανουάριο. Θα ήθελα να ζητήσω τώρα την κυρία Μπιόρκ να μας κάνει μια σύντομη παρουσίαση της κατάστασης των πραγμάτων. Κυρία Μπιόρκα, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαι όντως πολύ σύντομη. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Κιώδης που ενεργά συμμετείχαν ε, στους τριμερείς διαλόγους. Είχαμε μια πρώτη, ε, ένα πρώτο τριμερί πριν το τέλος του έτους με την Εστονική Προεδρία και καταλήξαμε σε κάποιες γενικές θέσεις ε, και μετά είχαμε και τον πρώτο διάλογο με ουσιαστική συζήτηση με την Βουλγαρική Προεδρία την 17η Ιανουαρίου. Όπως εξήγησε και η Σοφή προηγουμένως, ήταν σαφές ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές ανάμεσα στις δικές μας θέσεις και την, ε, ε, την ε, εντολή που έχω όσον αφορά το Κοινοβούλιο σχετικά με την εγκατάσταση, την ανθρωπιστική υποδοχή. Αυτό είναι ένα ευαίσθητο θέμα, θα το συζητήσουμε στον δεύτερο τριμερί συζητήσαμε για το πεδίο εφαρμογής ε, της ε, ανθρωπιστικής ε, υποδοχής. Πάντως χρήζει περαιτέρω συζητήσεως το θέμα έτσι ώστε να δούμε που θα ταυτιστούν οι θέσεις των ε, συνομοθετών. Επίσης, συζητήσαμε και τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Και εδώ υπάρχουν διαφορές ε, ουσίας ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδιαίτερος δε όσον αφορά ε, την, τις αρχές μη επιλεξιμότητας. Ε, πάντως υπάρχει η πρόθεση περαιτέρω συζήτησης έτσι ώστε να βρούμε κάποιους κοινού τόπους. Ε, προσδοκώ λοιπόν ε, σε, μια τρίτη, σε ένα τρίτο τριμερή διάλογο και καταγράφω την καλή στάση και καλό κλίμα από πλευράς Βουλγαρικής Προεδρίας. Επίσης, να υπογραμμίσω ότι είναι ανάγκη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να έρθει στην συζήτηση με συμβαστικές τροπολογίες οι οποίες ε, θα συγκλίνουν τις δύο διαφορετικές θέσεις ε, στη διάρκεια της διαδικασίας. Και αν τα καταφέρουμε αυτά πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να προχωρήσει ως global player σε μια στιγμή δηλαδή που είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε την ιδέα ότι προχωρούμε ε, κοιτάξτε, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που ακούσαμε. Εγώ θα ήθελα ε, να μάθουμε και περισσότερες ε, πληροφορίες. Δηλαδή, ποια είναι τα κύρια... Πότε είχατε κάποιο πρόβλημα τεχνικό. Okay. Can I try? Um, να τα ξαναπώ λοιπόν. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, θεμελιώδου σημασία και θα πρέπει να το συζητήσουμε. Πρόκειται για ένα θέμα απολύτω ευαίσθητο, κυρίω πριν τι εκλογέ. Γιατί ήταν και κεντρικό θέμα των ε, προηγουμένων εκλογών. Και ο πρόεδρο ο οποίο κέρδισε τι εκλογέ σε εμά ήταν αυτό ο οποίο μίλησε ακριβώ για την μετανάστευση. Και επομένω είναι θεμελιώδου σημασία. Θα πρέπει να δούμε με τι ε, επιπίων θεμάτων συμφωνούμε και τι, με τι διαφωνούμε. Ε, Ωραία. Και λέει κυρία Μπόρκο, ευχαριστώ πολύ να κάνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να αναλάβει περισσότερες ε, και πιο συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Το Συμβούλιο είναι πολλά, μπορούμε να τα συζητήσουμε αν θέλετε και διμερώς και οπωσδήποτε οι σκιώδεις συζητούν τις δυνατότητες εξέβρεσης συμβιβαστικών. Σοφή Ιντβελτ, θέλεις όχι να ξεκινήσουμε συζήτηση τώρα, μα πάρα πολύ ευαίσθητο όσον αφορά τη, τα εσωτερικά πολιτικά ζητήματα των χωρών. Έτσι όπως το βλέπω εγώ τουλάχιστον, η θέση του Συμβουλίου ή στην πράξη τι μπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα ή τι μπορεί να λειτουργήσει πραγματικά. Εγώ πιστεύω και αυτή είναι και θέση νομίζω του συνόλου της του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της σε πολλές χώρες. Αυτό είναι αλήθεια. ευχαριστώ πολύ. Φτάνουμε στο επόμενο και τελευταίο σημείο της σημερινής συνεδρίασης, πλουραλισμό στα μέσα ενημέρωσης και ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, η κυρία Σπινέλη. Παρουσίασε την έκθεσή της στις 11 Ιανουαρίου. 227 τροπολογίες έχουν κατατεθεί στην έκθεση Σπινέλη. Θα της δώσω το λόγο για να σχολιάσει τις τροπολογίες και τα θέματα που έθεσαν οι συνάδελφοι για μια τόσο σημαντική έκθεση. Κυρία Σπινέλη, το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω καταρχάς τους κοιόδης για τις τροπολογίες τους Κάθε μία από αυτές περιλαμβάνει πολύ σημαντικά στοιχεία και πολλές καλές προτάσεις που θέλουν να βάλουν στο κείμενο νέα καινοτόμα στοιχεία. Και νομίζω ότι οι επόμενες συναντήσεις προτάσεις που θέλουν να βάλουν στο κείμενο νέα καινοτόμα στοιχεία και νομίζω ότι οι επόμενες συναντήσεις των σκιωδών θα είναι στιγμές παραγωγικές ε, διαλόγου. Προκατακτικά λοιπόν πω αυτά τα οποία προτείνω εγώ σαν εισηγήτρια και αυτά τα οποία εγώ θεωρώ σημαντικά. Δεν θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να δώσουμε οδηγίες σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε από τις παραδοσιακές εφημερίδες, τα blog, να τους πούμε να λένε ή να μην λένε την αλήθεια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μία ερμηνεία των πραγματικών γεγονότων και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι τα μέσα ενημέρωσης είναι ένα μαντίο των δελφών που αναφέρονται σε θέματα με ενεργματικό τρόπο και αφήνουν τον αναγνώστη ακροατή να καταλάβει το νόημά τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο μόνο σε ολοκληρωτικά καθεστώτα μπορεί να σταθεί. Εμάς λοιπόν ο ρόλος μας δεν είναι διακανονιστικός αλλά πολιτικός και η πολιτική σύμφωνα με μένα στο Κοινοβούλιο σημαίνει ότι θα πρέπει να επιμείνουμε στην πίστη μας, στον πλουραλισμό, στην δημοκρατία και στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης που υπόεφεραν από τις ε, οικονομικές κρίσεις. Και θέλουμε τα μέσα ενημέρωσης να παραμείνουν η τέταρτη εξουσία ανεξάρτητες από άλλες μορφές εξουσίας όπως της πολιτικής και της δικής μας στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο ρόλος αυτής της τέταρτης εξουσίας είναι η κριτική λοιπόν εγώ αναφέρομαι σε αυτά τα οποία έχει πει για την κριτική ο Μισελ Φουκό. Είπε ότι η κριτική είναι η τέχνη που ασκούν οι κυβερνώντες έτσι ώστε να μην κυβερνηθούν με τη σειρά τους ποτέ. Δεν αγνοούμε εμείς στο ψήφισμα ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, το πρόβλημα των fake news πάνω στα οποία κατατέθησαν πολλές τροπολογίες. Η γνώμη μου είναι γνωστή. Την είπα εδώ στη Λίμπε και την επαναλαμβάνω και στην έκθεση. Δεν νομίζω ότι τα fake news είναι ένα νέο φαινόμενο και δεν νομίζω ότι μπορούμε να αντισυνδέσουμε συνδέσουμε μόνο με την έλευση του ίντερνετ και των κοινωνικών δικτύων. Θυμίζω εδώ τον πόλεμο στο Ιράκ και τις αναλήθειες που είχαν κυκλοφορήσει για τα όπλα μαζικής καταστροφής. Όλοι οι πόλεμοι που έκαναν οι Ηνωμένε Πολιτείε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με ή χωρίς την Ευρώπη μεταφέρθηκαν με στρεβλό τρόπο από παραδοσιακά μέσα με δημοσιογράφους οι οποίοι υποτίθεται ήταν ενσωματωμένοι στις πολιτικές, ε, στις στρατιωτικές δυνάμεις. Και υπάρχουν πολλές τροπολογίες που επιβεβαιώνουν την άποψή μου αυτή. Θα ήθελα λοιπόν το έγγραφο αυτό να έχει πάντα σαν, προσοχή, σαν κεντρικό θέμα τον πλουραλισμό και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και να μην γίνει ένα μέσο για να αντιμετωπίσουμε εγκάρσια θέματα τα οποία έχουν ήδη αντιμετωπιστεί από το Κοινοβούλιο αυτό σε άλλα ψηφίσματα όπως η καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή η πρόληψη της βίαιης των βίαιων ακραίων πολιτικών. Ένα άλλο θέμα είναι η αναφορά στην Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στον μηχανισμό τον οποίο προτείνει η Ιντβελτ για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, στα θέματα της δίωξης των ανεξαρτήτων δημοσιογράφων, στην αυτολογοκρισία, στην προστασία των ε, μαρτύρων ε, κοινή ωφέλεια σε εισαγωγικά. Όλα αυτά είναι διεθνικά θέματα. Αναφέρεται στα θέματα αυτά το ψήφισμα και μεταφέρει συγκεκριμένα αιτήματα για αυτά του Κοινοβουλίου. Στα πλαίσια λοιπόν αυτών των νέων και ανεξάρτητων μηχανισμών για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά διατυπώνεται μέσα από τροπολογίες που κατέθεσα και εγώ έτσι ώστε να, ενσωματίσουμε, να ενσωματώσουμε συγγνώμη, ότι για λόγους χώρου, χωρητικότητας δεν υπάρχει στην αρχική πρόταση. Υπάρχουν και άλλα θέματα που μέσω των νέων τροπολογιών η ουδετερότητα του δικτύου σαν παράδειγμα μετά από την απόφαση των, της Επιτροπής Μεταφορών και Επικοινωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών, η καθιέρωση των κανόνων για τη λειτουργία μέσω των διεθνών οργανισμών, η προώθηση του ψηφιακού αλφαβητισμού σε εισαγωγικά πάντα, και επίσης ο βασικός ρόλος που έχει να παίξει ο δημόσιος τομέας έτσι ώστε να δοθούν οι μέγιστες δυνατές εγγυήσεις από τις ομάδες πίεσης σε πολιτικό ή οικονομικό ή άλλης φύσεως επίπεδο. Υπάρχουν επίσης οι νομοθετικές ρυθμίσεις για την συκοφαντία, κάτι το οποίο θα πρέπει να επανεξεταστεί γιατί πολλές φορές έχουν σαν μορφή την, σαν στόχο την προστασία των πολιτικών και την ποινικοποίηση της δημοσιογραφικής δραστηριότητας. Δεν θα πρέπει με νέα μέτρα να λάβουμε να στραφούμε εναντίον της οικοφαντικής δυσφήμισης αλλά να πάρουμε σε αστικό επίπεδο μέτρα τα οποία να επιτρέπουν τον έλεγχο τους. Τώρα για την ρητορική μίσους ε, μετά από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2016 νομίζω ότι εκεί υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Υπάρχει ένα ιδιαίτερα μεγάλο περιθώριο διακριτικό στους ε, μεγάλους ε, του ίντερνετ όπως Facebook, YouTube, Google κτλ. Και κλείνοντας θα ήθελα να πω στους Κιώδης ότι η συνεισφορά τους θα είναι πολύ σημαντική, θα αναζητηθούν και ήδη έχουν ξεκινήσει να αναζητούνται συμβιβαστικές προτάσεις από χθε. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα ο κύριος ε, Μέλο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα ε, να πω ότι δεν θέλω να μπω τώρα σε αυτές τις λεπτομέρειες που μας παρουσίασε η κυρία Σπινέλη. Δεν θα τις ε, δω στο μικροσκόπιο. Πρέπει να σας πω ότι εγώ διαφωνώ με την εισηγήτρια. Και ακόμα και ενοιολογικά. Εγώ πιστεύω σε μια κοινωνία αξιών δεν ε, υποστηρίζω διάφορα ε, κινήματα. Ζούμε σε ένα κράτος δικαίωση δια του τύπου. Αυτή είναι μια κλασική περίπτωση χαρακτηριστική τα οποία ε, τα συζητούν και τα, στα πανεπιστήμια, στις σχολές δημοσιογραφίας. Υπάρχει το δικαίωμα στην ενημέρωση βεβαίως, για το αφισβητώ, αλλά υπάρχει και το δικαίωμα στην τιμή, στην αξιοπρέπεια και στο καθβάλι τον κόσμο χρησιμοποιώντας πολύ συχνά ένα πάρα πολύ ισχυρό οπλοστάσιο γιατί έχουν ε, πολλούς αναγνώστες, πολλούς ακροατές, πολλούς που τους ακολουθούν στα social media. Αυτό θίγει αξιοπρέπειες και που θα πρέπει να διέπεται και να πλαισιώνεται από αρχές και αξίες. Βεβαίως δεν είναι πάντα μία η εκδοχή της αλήθειας. Μπορεί ο καθένας να έχει τη δική του αλήθεια, αλλά δεν θα πρέπει κανείς προμελετημένα και εσκεμένα να αποσκοπεί στο να βλάψει ένα άλλο. Ε, έχουν ζωή και μέλλον. Εγώ προέρχομαι από μία νοτιοευρωπαϊκή χώρα όπου η φήμη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί κάποιοι αυτοί να το θεωρούν δευτερεύον στη Βόρεια Ευρώπη. Και υπάρχουν και καλοί και κακοί δημοσιογράφοι και καλόπιστοι και κακόπιστοι και επαγγελματίες και πολλά στη δημοσιογραφία. Υπάρχουν και κάποιοι δημοσιογράφοι λοιπόν που θεωρούν ότι έτσι ανυπόλογοι και να λογοδοτούν στη δικαιοσύνη. Για το λόγο αυτό δεν μπορώ να συμφωνήσω όταν γίνεται λόγος για αυτή τη σύγκρουση που υπάρχει για το αν είναι αξιόπινη πράξη η συκοφαντική δημοσιεύματα και ρίχνει λάσπη σε μένα, στην οικογένειά μου και ένα σπηλώσει το όνομά μου, αυτό θα πρέπει κάπου να λογοδοτεί. Και αυτό ο δημοσιογράφος πρόσωπο είναι. Δεν είναι κάτι το απρόσωπο. Όταν κάποιος μου επιτεθεί, όλοι οι πολίτες είναι ίσοι έναντι του νόμου. Δεν πάνε να είναι και δημοσιογράφοι, μάγειρες, πρόεδροι της δημοκρατίας. Ε, εάν ε, παραβαίνει το νόμο ένας δημοσιογράφος θα πρέπει να λογοδοτεί. Θα έρθω λίγο τώρα και στη αμπέλια όπου επιτρέπονται τα πάντα. Στην καθημερινή μα ζωή εμεί οφείλουμε να υπακούμε σε κάποιους κανόνες. Και όταν γίνονται σχόλια στο διαδίκτυο και ακούγονται διάφορες απόψεις η διασπορά ψευδών ειδήσεων δεν μπορεί να επιτρέπεται για να υπονομεύει την κοινωνία. Αυτό είναι αναρχία. Πρέπει να απαγορεύονται αυτά τα πράγματα. Και θα πρέπει να αποσκοπούμε όλοι στο να οικοδομήσουμε μια καλύτερη κοινωνία. Και οι μάρτυρες ε, δημοσίου συμφέροντος, οι whistleblowers, έχουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν. Δεν το αφισβητώ καθόλου. Ποιο είναι το καθεστώς αυτόν, το προστατεύονται αυτοί οι μάρτυρες. Όταν όμως κάποιος συνειδητά διασπείρει ψευδείς ειδήσει, ξέρει ότι ψεύδεται, τι προστασία να του ε, εξασφαλίσεις και πώς θα τον εντάξεις στο καθεστώς του προστατευόμενου μάρτυρα. Προστατεύεσαι και από πάνω. Αυτά είναι κατά χρήση του συστήματος. Δεν μπορείς να προστατεύεις τον εγκληματία. Για να ρίξουν λάσπη. Αυτά, λίγα μόνο ε, πρώτα σχόλια. Έχω πάρα πολλά ακόμα και τροπολογίες να κάνω. Απλώς ήθελα να σας αναφέρω αυτά σημαντικά για μένα. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Καταρίνα. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα πρώτα απ' όλα βεβαίως να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Σπινέλη ε, για την εργασία που έχει κάνει μέχρι τώρα και για, το, για τη μελλοντική της εργασία αυτή που θα κάνει μαζί βέβαια με τους σκιώδεις συγητές. Την ευχαριστώ για τις πολλές τροπολογίες που έχουν ε, υποβληθεί και που ε, αφορούν πολλά θέματα τα οποία εγγράφονται στην έκθεση. Πολλά θέματα αφορούν ε, περίπλοκες, ε, περίπλοκα στοιχεία και καταστάσεις που είτε εμπλέκονται μεταξύ τους είτε είναι εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους. Ε, Πρόκειται για μια έκθεση ιδιαίτερα ε, ε, ευαίσθητη ε, γιατί υπογραμμίζει στοιχεία τα οποία επανειλημμένα έχουμε συζητήσει εδώ, δηλαδή το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης και την προστασία του δικαιώματος αυτού, αλλά και την προστασία της ανθρώπινης ασφάλειας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζονται και στις ε, τροπολογίες ε, και στους ε, συμβιβασμούς που είναι πολυπληθείς και από τον οποίο θα πρέπει να εργαστούμε. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι το θέμα της συγκέντρωσης μέσων, οι ψευδείς ειδήσει, οι διατάξεις οι οποίες αφορούν τη μείωση της εξάρτησης των μέσων ενημέρωσης από την από την διαφήμιση, το, η ισότητα των φύλων, ε, κατά την άποψή μου αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Έχω υποβάλει και εγώ τροπολογίες ε, για το θέμα της προστασίας ε, των καταγγελόντων, των whistleblowers γνωρίζουμε ότι οι καταγγέλλοντες μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος και επομένως ε, θα πρέπει να έχουμε μια γενική τοποθέτηση η οποία ε, θα έχει σαν γενικό προσανατολισμό την προστασία ε, εξίσου σημαντικές οι αρχές και προστασίας των ε, ε, ανηλίκων, αναφέρομαι κυρίως στον κυβερνοεκφοβισμό, cyberbullying που, έχουν, ε, εποχή θύματα ανηλίκους. Ε, επίσης, ε, προσοχή και έλεγχος με ταυτόχρονη και άμεση παρέμβαση των εμπλεκομένων φορέων έτσι ώστε να αποκαλύπτονται γρήγορα τα περιεχόμενα συνομιλιών κλπ. Επίσης, οτιδήποτε αφορά αφήγημα μύθου, μίσους, ε, hate speech κλπ. θα πρέπει να μας απασχολήσουν ιδιαίτερως, γιατί πρόκειται για θέματα ε, ευαίσθητα και ιδιαίτερα περίπλοκα. Για όλα αυτά τα ευαίσθητα και περίπλοκα θέματα πιστεύω ότι ε, θα πρέπει να υπάρξει ε, η συνεργασία των ε, ε, ιδιωτικών μέσων, facebook, twitter κλπ. Και οπωσδήποτε όμως θα πρέπει οπωσδήποτε να αξιολογείται και η δυνατότητα αφαίρεσης περιεχομένου από το διαδίκτυο που θα πρέπει να ακολουθεί και να διέπεται από συγκεκριμένους και ξεκάθαρους κανόνες και γραμμές ε, ε, προσανατολισμού. Ξέρουμε ότι πολλά θέματα περνούν μέσα από τα μέσα ενημέρωσης. Επομένως, από τη μία πλευρά θα πρέπει να σεβαστούμε την ελευθερία έκφρασης, από την άλλη όμως θα πρέπει να διασφαλίσουμε την αξιοπρέπεια και την ασφάλεια των πολιτών. Επίσης υπάρχουν και θέματα ε, τα οποία είναι ιδιαίτερα περίπλοκα. Ε, αναφέρθηκε ήδη προηγουμένως ο συνάδελφος αυτό το της συκοφαντίας. Επ' αυτού πιστεύω ότι θα πρέπει ο καθένας μας ε, να το σκεφτεί, να το μελετήσει και ευελπιστώ ότι η συζήτηση μεταξύ των σκιωδών επί των συμβαστικών τροπολογιών. Ευελπιστώ λέγω η συζήτηση ολοκληρώσουμε να ξεκαθαρίσουμε ε, την ε, έκθεση ε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ε, προστατεύσουμε την ελευθερία της έκφρασης που αποτελεί πυλώνα της δημοκρατίας αλλά ταυτόχρονα να μην ε, καταπατηθούν δικαιώματα των πολιτών. Οπωσδήποτε να αντιμετωπιστούν. Να προβλέψουμε λοιπόν και κάποιες παρεμβάσεις εκπαιδευτικού ε, περιεχομένου και αξίας. Ε, οπωσδήποτε εμείς θα πρέπει να αξιολογήσουμε ε, τις ενδείξεις και θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε πάνω στο έγγραφο. Αυτό ευχαριστούμε πάρα πολύ την Μπάρμπαρα Σπινέλη για την εργασία που έκανε και ένα καλό συμβιβασμό. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ Κατερίνα. Ο κύριος Γιούρεκ, σκιώδης των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα πω κάτι που έχω επαναλάβει και στο παρελθόν. Εμένα μου αρέσει ως προπετούμενο για τη δημόσια συζήτηση έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί σωστά μια κοινωνία. Και να υπάρχει και δημόσια ευθύνη και λογοδοσία. Είναι καλή αυτή η προοπτική. Λυπάμαι όμως που στις συμβαστικές τροπολογίες λείπουν κάποια πράγματα. Άλογος δημόσιος να οικονομηθεί από την αρχή. σε κοινωνίες που είχαν γνωρίσει ολοκληρωτικά καθεστώτα και που δεν υπήρχε τέτοιος διάλογος. Σε περιπτώσεις που κλείνουν εφημερίδες, που υπήρχαν καταλήψεις σε μέσα ενημέρωσης, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Υπάρχει πρόβλημα και θα πρέπει να το λύσουμε. Υπάρχουν κάποιες κοινωνίες και κάποιε κάποιες ομάδες στην κοινωνία που κατά τη διάρκεια του ολοκληρωτισμού είχαν περιθωροποιηθεί. Πολύ συχνά το Η διάρκεια της μετάβασης στη δημοκρατία ε, συνεχίζουν τις διακρίσεις απέναντι σε εκείνους που τους θεωρούν δημόσιους εχθρούς και τους έχουν στιγματίσει. Θα πρέπει να μας προβληματίσει αυτό. Ή να μην έχει λόγο Αυτά τα θέματα εμείς τα είχαμε θίξει στις δικές μας τροπολογίες και παρακαλώ να ληφθούν υπόψη. Στη συνέχεια έχουμε το ζήτημα της λογοκρισίας και πάλι το τονίσαμε εμείς στις τροπολογίες μας. Υπάρχουν αυτό είναι αντίθετο με τις βασικές μας αρχές. Παράδειγμα, θυμάστε τον πόλεμο του Βιετνάμ. Ε, θυμάστε, οπότε οι εικόνες, οι τηλεοπτικές τον παρουσίαζαν ήρωα. Ε, πρέπει να έχουμε δικαίωμα στην αλήθεια. Για να συμμετέχουμε στο δημόσιο λόγο, γνώμονας θα πρέπει να είναι η αναζήτηση της αλήθειας. Ε, θα πρέπει να υπάρχει και μια αίσθηση της δεοντολογίας, της ηθικής. Τα λέμε στις δικές μας τροπολογίες επίσης. Άλλο θέμα